Παρακαλώ πολύ, καθίστε για να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. We have a vote. Έχουμε ψηφοφορία σε λίγα λεπτά. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διαταξής μας είναι η έγκριση αυτής. Το σημείο 18, η έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών ε, της Επιτροπής μας θα αναβληθεί για τον Ιανουάριο και αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη, τότε μπορεί να εγκριθεί. Επόμενο σημείο, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 12 Νοεμβρίου του 2015. Και αυτό θα αναβληθεί για τον Ιανουάριο γιατί δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι μεταφράσεις. Θα ήθελα εκ μέρους της Προέδρου να σας ενημερώσω ότι στη γραμματεία μας ε, έχουμε μία νέα βοηθό. Δεν είναι όμως εδώ. Μανών Μπόρμα λέγεται. Είναι Όλανδη. Όταν θα έρθει θα μπορέσει να μας συστηθεί. Θα θέλαμε πάντως ε, να την καλωσορίσουμε. Έχει εργαστεί σε άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς ε, και είμαι βέβαιη, ότι θα την καλωσορίσετε και θα τη βοηθήσετε όλοι σας. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχουμε δύο ψηφοφορίες. Η μία αφορά την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2014 θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η κυρία ε, κύριος Γκέριγκερ θέλει το, ε, το λόγο ή κυρία Γκέριγκερ, συγγνώμη ε, και θα ήθελα να σας πω ότι πρώτη φορά προεδρεύω ψηφοφορίας ε, και να σας ζητήσω να είστε ποιικείς μαζί μου. Κυρία Γκέριγκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, και τους συμβούλους. Λειτουργεί τώρα η διερμηνία στα αγγλικά. Ναι, λειτουργεί η διερμηνία. Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Όπως έλεγα λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κοιόδης εισηγητές ε, και τους συμβούλους μας, διότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά, δεδομένου ότι ήταν και πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι η έκθεση δραστηριοτήτων μας για το 2014, όταν ε, η Επιτροπή Αναφορών ασχολήθηκε για τρεις μήνες με το θέμα αυτό, θα είχε τόσα προβλήματα. Ε, και τελικά ε, είχαμε 180 ε, τροπολογίες ε, και μία συζήτηση που ορισμένες φορές ήταν και περιττή. Ε, χαίρομαι όμως που καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα και ελπίζω ότι οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση και οι συζητήσεις που έγιναν εδώ στην Επιτροπή προσέδωσαν τη δέουσα σημασία στην έκθεση και είναι μια έκθεση που είναι καλύτερη από αυτή που είχαμε στην αρχή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία για τα όσα έκανε και για την υπομονή της. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Hans Becker, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. να σχολιάσω και τις διαπιστώσεις της ε, εισηγήτριας. Μίλησα για ένα εκτενές έργο τριών μηνών. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η δουλειά έγινε αποκλείοντας πλήρως το ΕΛΚΑ από την εργασία της Επιτροπής αυτής ε, αναφορών. Είναι απαράδεκτο και θα ήθελα λοιπόν να σας πω ε, και να σας εξηγήσω γιατί αναγκαστικά θα απορρίψουμε την έκθεση αυτή. Καταρχάς, η διαδικασία απαράδεκτη. Δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της ψηφοφορίας, προχθές έγινε η πρώτη συνάντηση σκιωδών. Είναι πραγματικά απαράδεκτο και δεν αποτυπώνει φυσικά το χαρακτήρα και τη σύνθεση της ε, Επιτροπής. Πρόκειται για μια έκθεση ε, για την έκθεση 14-13, όπου εκεί αποτυπωνόταν η άποψη της Επιτροπής ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα email, τίποτα. Αυτό είναι πραγματικά άνω ποταμών. Και κανείς από τους ε, βουλευτές της ομάδας ε, δεν μπορεί να συμφωνήσει. Από τις 40 τροπολογίες, μόνο 5 συμπεριλήφθησαν του ΕΛΚΑ. Και καταλαβαίνετε, αυτό είναι σκόπιμο. Δεν υπήρξε καμία διάθεση για να υπάρξει μια συνέχεια σε ό,τι αφορά την προηγούμενη υποστήριξη που ήταν ευρεία. Επίσης, όλα τα βασικά κριτήρια τα οποία είχαμε ορίσει εδώ, είχαμε ορίσει για παράδειγμα ότι χρειαζόμαστε ναι, γρήγορη δουλειά, είχαμε ορίσει τις προθεσμίες, είχαμε συμφωνήσει ένα νέο σχέδιο με τη γραμματεία. Όλα αυτά δεν τρίθηκαν. Και δυστυχώς, δυστυχώς λέω, η ALDE και το ECR δεν τα ακολούθησαν αυτά. Και οι υπόλοιπε ομάδε. Κοίταξαν και τις, ε, τις συναντήσεις των σκιωδών ξεχωριστά. Νομίζω ότι είναι σαφές. Ε. Και υπάρχει μία άρνηση εκεί που έγινε τα συμφέροντα των ε, αναφερόντων. Εκεί δηλαδή που έχουν πραγματικές επιθυμίες και ανάγκες για επιτάχυνση των διαδικασιών οι πολίτες για τα κριτήρια αυτά. Όλα λοιπόν αυτά ήθελα να τα έχω αναφέρει προκειμένου να γνωρίζετε ότι είναι πραγματικά αδύνατον να δεχτούμε και να επιδοκιμάσουμε μια τέτοιου είδους ε, συνεργασία. Και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που εσείς αναλάβατε αυτή την έκθεση και με τον τρόπο αυτό Ε, συνεχίζεται έτσι αυτή η έκθεση η οποία είχε την υποστήριξη της Επιτροπής εδώ και χρόνια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πήξα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέρινγκ, να δώσω το λόγο στον κύριο Μαριά και μετά στην κυρία Βεσέρα. Κυρία Μαριά. Ε, κυρία Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο γιατί ήρθαμε για να ψηφίσουμε με μια διαδικασία ψηφοφορίας και ο καθένας είχε τη δυνατότητα και κάθε πολιτική ομάδα να εκφράσει τις απόψεις της και βεβαίως να εκφραστεί τώρα και δια της ψήφου. Επειδή όμως ο συνάδελφο αναφέρθηκε στο ECR, εγώ θέλω να πω ότι συμμετείχαμε με καλόπιστο τρόπο στις διαδικασίες των Shadows και συναντήσαμε ε, θα έλεγα ένα θετικό κλίμα από πλευράς της συγκήτριας. Οι απόψεις μας τέθηκαν, άλλες έγιναν δεκτές, άλλες δεν έγιναν. Από εκεί και πέρα είναι η ώρα της ψηφοφορίας. Πάντοτε θα υπάρχουν μειοψηφίε και πλειοψηφίε. Συμβαίνει μερικέ φορέ μερικοί που είναι στην πλειοψηφία να βρεθούν καμιά φορά και στη μειοψηφία. Αλλά έτσι είναι η δημοκρατία και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία και να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Madame Becerra. Go ahead. Muchas gracias, Presidenta. Κυρία Βεσέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μαριά. Ούτε κι εγώ είχα σκοπό να λάβω το λόγο και νομίζω ότι η ευελιξία και ο ανοιχτό χαρακτήρας είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα μέλη της Επιτροπής των Αναφορών και πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο και στις προθεσμίε που έχουμε και να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στους πολίτες. Σε καμία περίπτωση οι πολίτες ε, και δι αναφέροντες δεν, ε, ε, που μας διαβιβάζουν τις αναφορές τους και τις καταγγελίες τους δεν φαντάζονται ότι δεν είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε και να συμφωνήσουμε για την έκθεση για τις δικέ μας τι δραστηριότητες. Νομίζω ότι δεν περιμένουν κάτι τέτοιο από εμά και σε καμία περίπτωση δεν περιμένουν να μπλεκόμαστε σε συζητήσεις και σε άνε δικαιολογίε και ατέρμονες συζητήσεις ε, και όπως είπε και ο κύριος Μαριάς, επιμένω και εγώ από πλευράς φιλελευθέρων η συζήτηση ήταν ανοιχτή, κάποιος προτείνει τις τροπολογίες του, γίνονται δεκτές, απορρίπτονται, αλλά ο κοινό στόχος είναι να έχουμε μία έκθεση που θα εξηγεί τις δραστηριότητες αυτής της Επιτροπής Αναφορών και να επενθυμίσουμε ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρονιά, το 2014, ε, έχουμε και νέα θητεία στο δεύτερο μισό του. Σε ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκέριγκερ, για να συνοψίσει και μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εκείνους που έλαβαν το λόγο. Πρέπει να πω ότι εκπλήσωμαι για αυτό που είπε ο κύριος Μπέκερ, διότι έγιναν δύο σημαντικές συζητήσεις ε, στη διάρκεια της συνεδρίας Επιτροπής Αναφορών. Εγώ πρότεινα να συναντηθούν νωρίτερα οι σκιώδεις εισηγητές ε, και πέραν του κυρίου Μπέκερ, ε, πέμπτη απόγευμα, κανείς δεν είχε χρόνο να συναντηθούμε και επομένως χρειάστηκε να αναβάλουμε τη συνεδρίαση για αργότερα. Έγινε ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ε, από πλευράς βοηθών μα, ίσως να μην λάβατε και εσεί τα μηνύματα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα να πούν την άποψή του και έτσι μπορέσαμε να καταλήξουμε και σε αυτέ τι συμβαστικέ λύσεις. Και εμένα με ικανοποιεί αυτό το αποτέλεσμα. Και πέραν από εσά δεν βλέπω κάποιον άλλον δυσαρεστημένο, δεν ξέρω ε, πόσες θέλετε εσεί να συναντιούνται οι σκιώδει εισηγητές αλλά εγώ θεώρησα ότι αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων και οι συζητήσει που έγιναν εδώ αρκούσαν. Από ό,τι φαίνεται για σας δεν αρκούν, για μένα όμως αρκούν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε επιτέλου στη ψηφοφορία. Λόγω του καταλόγου της ψηφοφορία που όπως βλέπετε περιλαμβάνει ένα αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών, παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Επιβεβαιώστε λοιπόν ότι η κάρτα σας είναι μέσα στο μηχάνημα. Και αρχίζω με την 81. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 82. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. 83. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Αγκρίνεται. 84. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 85. Έναρξη. Πέρας. Συμβιβαστική τροπολογία A. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. 92. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 93. Έναρξη. Είναι κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 94. Πέρας. Εγκρίνεται. Η Συμβασική Βήτα. Ενάρξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρα. Εγκρίνεται. Η 98 έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Η 99 έναρξη. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 100. Έναρξε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 101. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 102. Έναρξη. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Η 103. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 104. Καταπίπτει. Η 105 λέει η πρόεδρος. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Συ. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Ή 111 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται προφορική τροπολογία των πρασίνων να συμπεριληφθεί η λέξη well functioning μεταξύ create και addition. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 112. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 114. Ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία από τις πράσινες. Πρώτο τμήμα παρακαλώ έναρξη. Πέρας απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα τώρα, έναρξη. Πέρας. Και αυτό απορρίπτεται. 115. Σε τμήματα που έχει ζητήσει η Γκουε. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα παρακαλώ. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 116. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 117. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 118 έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 119. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έχει ζητήσει η δηλαδή. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 120. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 121. Έναρξη. Πέρας εγκρίνεται. Ή 123, 123, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 124 σε τμήματα μετά από αίτημα των πρασίνων το τμήμα έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 125. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 126. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 127. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 128. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 129. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας εγκρίνεται. 130 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D, δέλτα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 140, 138. Υπέρ. Μάλλον ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 139. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 140. ενέργεια, Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα. Περνάμε στην Okay, amendment 141, λέει η Πρόεδρος, ψηφίζουμε. Okay. Compatible with They don't fall because uh, this this is only if if if this is adopted and it was not adopted. It was it was adopted. Uh, Sorry. Sorry. Adopted. Amendment number one. 142 λέει η Πρόεδρος. Έναρξη. Έκλεισε ψηφοφορία για την 141 και λυπάμαι. Εγκρίνεται. 142 τώρα. Έναρξη. 142. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 143 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε προφορική γλωσσική τροπολογία των πρασίνων. Discrimination αντί για prohibition of discrimination. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 144. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε. Ή. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 150. Υπάρχει αίτημα ξεχωριστής ψηφοφορία από την ΚΟΕ. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία 151. Έναρξη. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 152. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 153. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 154. <coughs> Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 155 ή 156 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 157 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 158. Σε τμήματα μετά από έτοιμα της ΓΟΕ και των Πρασίνων. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 159. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 160. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 161. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 162. της η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 163. της η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβασική τροπολογία F. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ...168... Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία, εγκρίνεται. 169. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 170. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 174. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις παραθέσεις. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 7 καταπίπτει, τροπολογία 8, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ε, χωριστή ψήφος ε, κατά τμήματα ε, μετά από έτοιμα Τμήμα 1. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το τμήμα 2. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εκρίνεται. Τροπολογία 23. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Κατά τμήματα, ε, κατόπιν αιτήματο των πρασίνων, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 27, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30, η άρχεται ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 31, άρχεται ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, άρχεται ψηφοφορία. 37. Πέρας της ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας της φορείας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43, άρχεται ψηφοφορία, Πέρασε τη ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 44, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της Εγκρίνεται. Τροπολογία 45, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της Εγκρίνεται. Τροπολογία 46, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της Εγκρίνεται. Τροπολογία 47, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Άρχεται ψηφορία. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Άρχεται ψηφορία. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Άρχεται ψηφορία. Πέρας της ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία I, στην αιτιολογική σκέψη N. Συμβαστική τροπολογία I. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 61 πριν πάμε στην ε, ε, συμβαστική τροπολογία J και να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Welcome μέχρι savings. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στη συμβαστική τροπολογία J. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 71, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία, Εγκρίνεται. Τροπολογία 72, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. Τροπολογία 73, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία, Εγκρίνεται. Τροπολογία 74, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Να Τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και τώρα περνάμε στην τελική ψήφο για το σύνολο της έκθεσης άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 17 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Ωραία, σας ευχαριστώ και πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία για τις δύο προφορικές ερωτήσεις. Που θα είναι πολύ συντομότερη. Κοινή προφορική, προφορική ερώτηση ε, σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων των παιδιών διασυνοριακά στην Ευρώπη. Μία ψηφοφορία για την, ε, για την προφορική ερώτηση συνολικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 27 ψήφοι υπέρ και προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των καλύτερων συμφερόντων των παιδιών μία ψηφοφορία πριν περάσουμε στο σύνολο της ε, ερώτησης όλο το κείμενο εκτός από την αναφορά στις χώρες Γερμανία, Δανία ε, κλπ. Οπότε πρώτα ψηφίζουμε αυτό το τμήμα. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε την προσθήκη των χωρών στην παράγραφο 4, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Why did you vote of them? Okay, let's vote Λοιπόν, να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της ερώτησης, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίναμε την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 27 ψήφους υπέρ και καμία ψήφο κατά. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you everybody. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που ήταν εδώ για την ψηφοφορία. Να περάσουμε τώρα ε, στην ε, ε, υπόλοιπη ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Έχουμε δύο, τρεις αναφορές. Από τρεις Πορτογάλους αναφέροντες. για τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν τα σχολεία εκπαιδευτικούς στην Πορτογαλία που θεωρεί ότι αντιβαίνει στην ενωσιακή νομοθεσία γιατί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ε, εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παρακαλώ μήπως μπορείτε να κάνετε ησυχία, ειδικά όσοι φεύγετε. Μου λέει εδώ η γραμματεία ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Μισό λεπτό. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι ενό λεπτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Λοιπόν, αυτό που δεν είπα προηγουμένως είναι ότι είναι εδώ ο αναφέρον και αυτό που θα μας πει είναι ότι από τη στιγμή που υπήρξαν περιορισμοί στον προϋπολογισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, ε, ε, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος αναφέρον να έχει προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου επανειλημμένος. Τώρα έχουν ανοίξει διαδικασίες, εκεί οι διαδικασίες ε, επί παραβάση λόγω της παραβίασης οδηγίας 1999 και ε, στις 28 ε, Μαΐου κρίθηκε παραδεκτή η συγκεκριμένη αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παράβασης ε, γιατί Υπάρχει πλέον ένα όριο μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας σε πέντε χρόνια συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ANVPC είναι εδώ μαζί μας να μας παρουσιάσει την αναφορά του και του δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Καλημέρα σας. Ε, καλημέρα. Θα ήθελα να σας πω ότι παρουσιάσαμε ένα έγγραφο για την συνεδρίαση αυτή. Σας υποβάλαμε κάποιο έγγραφο, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τη μετάφραση εγκαίρω. Θα σας κάνω λοιπόν την παρουσίασή μου για την αναφορά μας που αφορά του συμβασιούχου καθηγητές. η κατάστασή μας ε, σίγουρα είναι λιγότερο ευνοϊκή από τους μονίμους ε, καθηγητές, το μόνιμο διδακτικό προσωπικό των ε, σχολείων στην Πορτογαλία για 7 λόγους. Καταρχάς για λόγους μισθοδοσίας. Οι αναπληρωτές και συμβασιούχοι καθηγητές έχουν ένα μισθό μειωμένο με μεγαλύτερο αριθμό διδακτικών ωρών ε, και λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν και λόγω ηλικίας. Ε, η πρόσληψη γίνεται σε αιτήσια βάση, ενώ οι μόνιμοι καθηγητές ε, φυσικά είναι έχουν περισσότερο χρόνο και γίνεται και αξιολόγηση μία φορά το χρόνο, ενώ για τους μονίμους καθηγητές προβλέπεται μεγαλύτερη ε, διάρκεια ανάμεσα σε δύο αξιολογήσεις. Και αν ένας καθηγητής ε, λάβει ε, ανεπαρκή βαθμό κατά την αξιολόγηση, για τρία χρόνια δεν μπορεί να προσληφθεί και δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση για πρόσληψη. Επίσης είναι πολύ σοβαρά κάποια πράγματα συγκριτικά γιατί κανένας συμβασιούχος καθηγητής δεν μπορεί να αποφύγει τη διαδικασία θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλει πιστοποιητικό καλής φυσικής και ψυχικής υγείας και πιστοποιητικό ποινικό μητρό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο ενώ δεν απαιτείται κάτι αντίστοιχο από το μόνιμο προσωπικό. Αυτά τα λέω για να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σας, διότι στην τελευταία ε, αξιολόγηση που έγινε το 2015 η μέση ηλικία ε, για μάλλον συγγνώμη, το μέσο διάστημα για το οποίο αποσχολούνταν κάποιος ήταν 13 χρόνια, ενώ υπάρχουν κάποιες ομάδες ε, που είναι στα 17 χρόνια υπηρεσίας. Για την ε, η πορτογαλική γλώσσα και για τα καλλιτεχνικά είναι 19 χρόνια και ε, επομένως όλοι όσοι έχουν 10, 15 χρόνια προϋπηρεσία, 20 χρόνια προϋπηρεσία δεν ε, προσλαμβάνονται άλλο, διότι το Πορτογαλικό κράτος ε, το 2014 πέρασε μια νέα νομοθεσία βάσει της οποίας τα πάντα βαίνουν καλό όσον αφορά του συμβασιούχου καθηγητέ. Ε, αυτό ήταν για να καθησυχάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ισχύει όμω κάτι τέτοιο, διότι βάσει πορτογαλική νομοθεσία ε, οι συμβασιούχοι καθηγητέ έπρεπε να έχουν πέντε συναπτά έτη, ένα συν τέσσερι ανανεώσει και έφτανε μία μέρα ε, αλλαγή ε, στη σύμβαση ή 30 συν μία μέρε και αυτό θεωρούνταν επαρκέ κριτήριο για να μην επαναπροσληφθούν. Και επομένως θα ξεκινούσε εκ νέου η διαδικασία και ξαναξεκινάει η προσμέτρηση αυτών των πέντε ετών προϋπηρεσίας. Ε, πρέπει να πω επίσης ότι οι συμβασιούχοι καθηγητές ε, έπρεπε να έχουν ετήσια σύμβαση από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 1η Αυγούστου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα, διότι η πρόσληψη γίνεται περιοδικά και το 2013 στις 15 Σεπτεμβρίου οι προσλήψεις έγιναν ε, ε, στις 15 Σεπτεμβρίου, φέτος έγιναν στις 12 Σεπτεμβρίου και επομένως η πορτογαλική κυβέρνηση θεώρησε ότι η έναρξη της σύμβασης ε, δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται από τη στιγμή πρόσληψης και θα πρέπει να ισχυσει αρνοαδρομικα αεροδρομικά από 1η Σεπτεμβρίου. Επειδή όμως ε, Λαμβάνεται υπόψη και η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ε, υπήρχε διαφορά από κάθε σχολική χρονιά στην άλλη και μάλιστα και από ένα σχολείο στο άλλο. Σε κάποια σχολεία ξεκινούσαν νωρίτερα και κάποια αργότερα. Κάποιοι λοιπόν καθηγητές και διδάσκοντες έχουν διαφορετικές ε, ημερομηνίες για την ε, ε, ημερομηνία πρόσληψή τους και επομένως η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Σας εξηγώ λοιπόν τα εξής. Η πορτογαλική νομοθεσία επιτρέπει τη διακοπή αυτών των διαδοχικών συμβάσεων και έτσι οι συμβασιούχοι καθηγητέ μπορεί να έχουν 10-15 χρόνια προϋπηρεσία... και βάσει αυτής της νομοθεσίας δεν μπορούν να έχουν 5 συνεχή έτη εργασία. Από την άλλη, η πορτογαλική κυβέρνηση τελικά άρχισε βάσει αυτή τη νομοθεσία να μετράει ω προπηρεσία μόνο την τελευταία πενταετία, από το 2010 μέχρι το 2015, ενώ οι περισσότεροι διδάσκοντες ε, στα 10-15 χρόνια που εργάζονται είχαν ε, ε, διαδοχικέ συμβάσει. Επειδή όμω προσμετρήθηκαν μόνο οι τελευταίε 5 χρονιέ, η τελευταία πενταετία και αυτοί βρίσκονται ζημιωμένοι. Επομένως, αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στην κινητική νομοθεσία για τις διαδοχικές συμβάσεις δεν ε, καλύπτεται εδώ διότι η πορτογαλική κυβέρνηση βρήκε έναν τρόπο να το παρακάμψει λέγοντας ότι έχει επιλύσει όλα τα προβλήματα ενώ στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν επιλύθηκε κανένα πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πολύ επισφαλής η θέση των συμβασιούχων διδασκόντων. Αυτό ισχύει για πολλούς συναδέλφους και επομένως θεωρούμε και σε αυτή την περίπτωση ότι επειδή η οδηγία προβλέπει ότι η Πορτογαλία όπως και όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πρέπει ε, να ε, βελτιώσει την ομοθεσία της ε, με βάση και την κοινοτική οδηγία, θεωρούμε ότι αυτό δεν έχει συμβεί και εξακολουθούμε να είμαστε σε πολύ επισφαλή κατάσταση. Υπάρχουν ακόμα λοιπόν συμβασιούχοι καθηγητές που έχουν 15 και πάνω περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας και ακόμα η κατάσταση αυτή διονύζεται και θεωρούνται ε, συμβασιούχοι που ξεκίνησαν την τελευταία πενταετία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Επιτροπή σας θα μπορέσει επιτέλους να λάβει μια απόφαση για να λάβει υπόψη τη την αναφορά μας, διότι θεωρούμε ότι γίνεται διάκριση εάν ε, ε, συγκρίνουμε την κατάσταση την οποία ζούμε εμείς σε σχέση με τους μόνιμους ε, καθηγητές. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι το βασικό προσωπικό οποιοδήποτε σχολικού ιδρύματος. Για μας λοιπόν ο ρόλος του διδάσκοντος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τα γαλλικά σχολεία και πρέπει να είναι ε, μια σταθερή κατάσταση. Θέλουμε λοιπόν να σταθεροποιήσουμε κάπως το λειτουργήμα που ασκούμε. Ολοκληρώνοντας κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Βρισκόμαστε σε πολύ επισφαλή θέση. Δεν έχουν δοθεί κατάλληλες απαντήσεις. Δεν έχει βρεθεί μια λύση για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στους κοινοκτικού κανόνες που έπρεπε να μεταφέρει η πορτογαλική νομοθεσία. Γι' αυτό άλλωστε ξεκίνησε και η διαδικασία επιπαραβάση. Και τελικά το πρόβλημα επιλύθηκε μόνο το 2014, αλλά εμείς ακόμα δεν έχουμε βιώσει κάποια σταθερότητα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα με χαρά θα δώσω τα λόγο στα μέλη της Επιτροπής, εν μάλλον στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Γκίν. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αναφέροντα, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, πράγματι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια με την αναφορά αυτή. Προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό γιατί έχουμε λάβει από το 2009 εκατοντάδες καταγγελίες για το θέμα αυτό. Αυτές οι καταγγελίες τότε αφορούσαν ε, την διαδοχή ε, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας για το την ίδια θέση και ειδικότερα σε σχέση με τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, ε, σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό και το θέμα της ε, αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ε, με το πέρασμα των χρόνων. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να υπενθυμίσουμε ποιες είναι οι βασικές διατάξεις της οδηγίας που αφορά τι συμβάσει ορισμένου χρόνου, μία οδηγία, σα υπενθυμίζω, που προέκυψε από συμβιβασμό μεταξύ των κοινωνικών εταίρων των επαγγελματιών του κλάδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τη ρήτρα 4, την περιβόητη, που αφορά τι συνθήκε εργασία. Πρόκειται για μία ρήτρα η οποία είναι μια ρήτρα ισότητας ε, ε, μεταχείρισης ε, Λέει λοιπόν ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να, τύχουν, να τυχαίνουν διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με τις του χρόνου, εκτός εάν δικαιολογείται για αντικειμενικούς λόγους. Επίσης, από την άλλη, υπάρχει η ρήτρα 5, η οποία είναι μια ρήτρα κατά της κατάχρησης που θα είχε ως ήταν αποτέλεσμα... Ε, ε, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση διαδοχικών συμβάσεων εργα, ε, εργα, εργασίας ορισμένου χρόνου. Τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να ε, συμπεριλάβουν στην ομοθεσία τους τουλάχιστον ένα από τα εξή μέτρα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα μέτρα που θα αναφέρω είναι σημαντικά, είναι απαραίτητα για να γίνει σεβαστή η ε, οδηγία. Πολλές φορές βέβαια γίνεται και ένα συνδυασμό των μέτρων αυτών, πάντως μία, ένα μέτρο αρκεί. Πρώτον, ε, αντικειμενικοί λόγοι που εξηγούν και δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ε, ορισμένου χρόνου διαδοχικά και ένας αριθμός ανανέωσης των συμβάσεων αυτών. Οπότε, σε γενικές γραμμές θεωρήσαμε ότι όντω υπήρχε παραβίαση τη οδηγία από πλευρά Πορτογαλίας όταν αρχίσαμε να ασχολούμε με το θέμα αυτό ε, και αρχίσαμε να ασχολούμαστε, να ερχόμαστε σε επαφή από το 2010 σε επαφή με τις πορτογαλικές αρχές. Θα ήθελα να πω το εξής όσον αφορά τη σχέση με τους καταγγέλλοντες ε, αναφέροντες που είναι παρόντες εδώ σήμερα ήρθαμε σε επαφή με τη ANPVC και λάβαμε πάντοτε υπόψη με πολύ προσοχή τις ε, πληροφορίες που μας είχαν ε, υποβάλει. Επίσης, κατόπιν αιτήματός τους ε, ήρθαμε σε επαφή με δύο Πορτογάλους συναδέλφους από την ομάδα Γκουε, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να έχει υπόψη της το ευρύτερο πλαίσιο της αναφοράς αυτής και πολλές φορές ε, ήρθαμε σε επαφή για δύο χρόνια με τις πορτογαλικές αρχές για να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα μπορούσαμε να ε, επιτύχουμε το στόχο μας. Τέσσερα στοιχεία συμπεριλαμβάνει η Πορτογαλική νομοθεσία σημαντικά. Πρώτον, η οργάνωση της ε, στρατηγικής πρόσληψης που δίνει τη δυνατότητα μόνιμης ε, πρόσληψης κάποιων εκπαιδευτικών, επίσης ε, διαδοχικών συμβάσεων πλήρους απασχόλησης πέντε ετών και τέσσερις ανανεώσεις. Τρίτον, αναγκαιότητα αντικειμενικών λόγων για την ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε δημόσιο αξίωμα και επίσης εμπειρία ε, που έχει αποκτήσει κανείς βάση συμβάσεων ορισμένου χρόνου που να μοιάζει με την εμπειρία ε, κάποιου συναδέλφου που έχει προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο περιθώριο στο πλαίσιο της νομοθεσίας αυτής. Ε, τα κράτη-μέλη όπως, όπως σας είπα προηγουμένως μπορεί να επιλέξουν ένα από τα μέτρα που ανέφερα. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας ε, πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν βάσει της νομοθεσίας του 2014 ε, και να εξασφαλίζουν την συμμόρφωση της Πορτογαλίας με την ενωσιακή νομοθεσία. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ομολογία του σε συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε ότι ε, δεν υπάρχει πρόβλημα με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου και τη συνεχή ανανέωσή τους αν κάθε φορά υπάρχει αιτιολόγηση με αντικειμενικούς λόγους. Βεβαίως το Δικαστήριο ζητά οι λόγοι αυτοί να ε, είναι πολύ συγκεκριμένη και σαφέστατη. Επίσης ε, υπενθύμησε ότι ε, είναι εναπόκειται στην εθνική δικαιοδοσία να επαληθεύει την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ε, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις. Το γεγονός ότι η πορτογαλική νομοθεσία περιορίζει στα πέντε χρόνια ε, ε, τη διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου είναι ένα επιπλέον, ένας επιπλέον περιορισμός και γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι μπορούμε να κλείσουμε τη διαδικασία επί παραβάση πριν από, μερικούς, πριν από μερικές εβδομάδες. Βεβαίως, λάβαμε πριν από μερικές εβδομάδες ε, από την ANVPC, δηλαδή από πλευράς του αναφέροντος, ε, ε, μακροσκελή ενημερωτικά έγγραφα που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτής της μεταρρύθμισης και αποφασίσαμε λόγω του μακροσκελούς χαρακτήρα να ε, ξεκινήσει και πάλι ε, μία διαδικασία. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη τις μεταφράσεις διαθέσιμες. Αν υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία ε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις πληροφορίες που λάβαμε. Και επί της βάσεως αυτής θα δούμε κατά πόσο πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις πορτογαλικές αρχές, αν υπάρχουν πραγματικά νέα δεδομένα σε σχέση με όλη την ομολογία του δικαστηρίου και την ερμηνεία της οδηγίας και του περιθωρίου ελιγμών που ε, υπάρχει για τα κράτη-μέλη. Και αν ισχύει αυτό, αν υπάρχουν νέα στοιχεία, θα έρθουμε σε επαφή με τις πορτογαλικές αρχές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ε, διαπιστώσουμε ότι η οδηγία έχει επιφέρει αποτελέσματα σε σχέση με την επισφάλεια των θέσεων εργασίας ε, στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες ε, τις συνδικαλιστικές, για παράδειγμα, κάποιων κρατών μελών και συγκεκριμένα, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η καταπολέμηση αυτού του αστικού θρύλου ότι η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ε, μετατρέψουν κάθε σύμβαση ορισμένου χρόνου σε μόνιμη σύμβαση. Δεν είναι αυτός ο στόχος της οδηγίας και το 2014 πολλές φορές ε, το υπενθύμησε αυτό το δικαστήριο. Ωστόσο, νομίζω ότι ε, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τη μεταρρύθμιση της πορτογαλικής νομοθεσίας χάρη στις καταγγελίες και στην αναφορά αυτή και θα ήθελα Ολοκληρώνοντας, να επενθυμίσω ότι οι διαδικασίες που ε, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν μόνο να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση του, της νομοθεσίας της Εθνικής Ενός Κράτους Μέλους με την Ενωσιακή Νομοθεσία και ε, υπάρχουν βέβαια και μεμονωμένες υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν καθαρά με την εθνική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, λεπτομερέστατη και συνεκτικότατη αυτή αναφορά στην Επιτροπή μας. Είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο αυτό. Και μας... Ε, και πολύ ενημερωτική. Μακάρι να τον είναι πάντα έτσι. Γιατί δεν είναι πάντα έτσι, ξέρετε. Εξαιρετική παρουσίαση. Να δώσουμε το λόγο στα μέλη της ε, Επιτροπής. Κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας καλωσορίσω να καλωσορίσω τον αναφέροντα ε, νόματο των ε, συμβασιούχων καθηγητών. Ακόμα και αν ε, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής σας, αποφάσισα να είμαι εδώ σήμερα το πρωί για να μπορέσω να επιβεβαιώσω τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Καθηγητών όσον αφορά την κατάσταση των συμβασιούχων καθηγητών στην Πορτογαλία. Ε, δεκαετίες ε, διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και πρέπει να πω ότι το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης ε, στην Πορτογαλία βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτές τις διαδοχικές συμβάσεις των διδασκόντων. Δηλαδή, το δημόσιο σχολικό σύστημα υπάρχει χάρη σε αυτού του συμβασιούχου καθηγητέ. Πρόκειται ούτω ή άλλω για επαγγελματίε, οι οποίοι έχουν προσφέρει ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν στη δημόσια εκπαίδευση με πολύ μεγάλε προσωπικέ οικογενειακέ θυσίε. Ορισμένε φορές είναι και μεγάλη αβεβαιότητα ε, για την ε, ε, βιωσιμότητά τους και το να μπορέσουν να έχουν και έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να τους ε, βοηθήσουμε. Πρέπει να πω επίσης ότι υπάρχουν διάφορα σωματεία καθηγητών και εξεγέρθηκαν ε, απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει συνέχεια στις συμβάσεις και μπορεί ορισμένες φορές ε, ε, επειδή ακριβώς ε, λύγει μια σύμφαση και υπάρχουν μια-δυο μέρες διακοπής οι αρχές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτό το παραθυράκι και να μην θεωρηθεί αυτή η διαδοχική σύμβαση. Πρόκειται για ένα σύστημα που βρήκε η κυβέρνηση για να μην σέβεται την ομοθεσία εν τέλει. Κατά την άποψή μας, η λύση θα ήταν να αλλάξει η νομοθεσία. Το έχουμε άλλωστε προτείνει στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ζητάμε να ληφθούν υπόψη οι μόνιμες ανάγκες των σχολείων και επίσης να γίνονται και προσλήψεις βάση του ωραρίου εργασίας ε, και να λαμβάνεται υπόψη και αυτή ε, η δυνατότητα διαδοχικής σύμβασης ουσιαστικά τιμωρούμε αυτούς τους καθηγητές. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ενέος κατάλογος, ο οποίος θα έχει και κατάλληλες διαβαθμίσεις φυσικά, ώστε οι καθηγητές ε, να μπορούν ε, να ε, τοποθετούνται στα διάφορα σχολεία, διότι πρόκειται για σχολεία που έχουν μόνιμες ανάγκες και προσλαμβάνουν συνεχώς τους ίδιους ανθρώπους. Επομένως δεν πρόκειται ε, δυστυχώς για μόνιμες θέσεις εργασίας και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Χωρίς όμως αυτούς τους καθηγητές δεν θα υπήρχε σχολείο. Δεν θα υπήρχαν δημόσια σχολεία στην Πορτογαλία αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καθηγητές. Εδώ και αρκετά χρόνια Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκε. Επομένως, θεωρώ ότι δεν με εκπλήσει και πάρα πολύ η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ορισμένες φορές ε, αντιδρά ταχύτερα και επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που δεν ε, ε, σέβονται μακροοικονομικούς κανόνες και πολύ συχνά είναι οι ίδιες χώρες οι οποίες στερούν δικαιώματα από πολίτες και λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε μία κοινωνική επιδείνωση σε αυτή την περίπτωση των εργατικών δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Δεν είμαι μέλο τη Επιτροπή σα, αλλά θέλω να κάνω δύο παρατηρήσει. Από ό,τι κατάλαβα από την παράβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η υπόθεση σήμερα άνοιξε ξανά. Σωστά κατάλαβα. Υπήρχε μια αναφορά η οποία είχε κλείσει και μετά Ε, χάρη στα επιχειρήματα και του αναφερομένου, ε, ξανά άνοιξε αυτή η αναφορά. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε και από πλευρά ε, διαδικασία που βρισκόμαστε. Και επίση, θα ήθελα να ρωτήσω και εσά ω μέλη τη Επιτροπή Αναφορά, αν κάποιο ξέρει να μου απαντήσει. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε εμεί εδώ στην Επιτροπή Αναφορών όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά. Η διαδικασία πώ έχει. Σα ευχαριστώ. Αυτή η αναφορά έχει μπει στην ατζέντα ε, μετά από αίτημα της ΓΚΟΕ. Θα... Πρέπει να πω λοιπόν ότι επέτρεψα στην ΓΚΟΕ να πάρει το λόγο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι επιτρεπόταν. 20 ε, λεπτά σχεδόν έχουμε αφιερώσει. Έχω τέσσερις ε, συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν, μιας και οι υπόλοιποι έχουν εξηγήσει τις, τα περιστατικά της υπόθεσης, να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Ο λόγος στον κύριο Μαρτά. Πραγματικά είστε πολύ αυστηρό μαζί μου. Ένα λεπτό μου δίνετε. Τι να πρωτοπώ σε ένα λεπτό. Θα το πω αυτό που έχω να πω και α πάρει λίγο παραπάνω. Να πω απλώς, ε, λόγω των εξηγήσεων που ακούσαμε, Προφανώ υπάρχει μια θέληση από πλευράς ε, πορτογαλικών αρχών ε, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί κατάλληλοι. Υπάρχει όμω η παραβίαση του υπερβολικού αριθμού ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ε, το, τη διαφορετική μεταχείριση των εκπαιδευτικών αναλόγως με τη σύμβασή του. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση αυτά που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν θέλω να πω τίποτε εναντίον της πορτογαλικής κυβέρνησης. Ε, απλώς, ε, εντάξει, δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απευθεία ένοχη, αλλά λέει στα κράτη-μέλη πρέπει να... Ε, να ε, σεβαστούν δύο ρήτρε ε, παρά το γεγονό ότι και οι ρήτρε αυτέ είναι εντελώ καταχρηστικέ. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά εφόσον υπάρχει νομολογία από πλευράς Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι, ότι όταν υπάρχει μία μόνιμη δραστηριότητα πρέπει να υπάρχει σύμβαση ε, αορίστου ε, χρόνου. Και θα το λέω αυτό ότι εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμάς μας έχουν καταδικάσει γιατί έχουμε κάνει τέτοιου είδους καταχρήσεις ε, των συμβασιούχων και κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί να ε, μπορέσουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω σε ποια δεδομένη χρονική στιγμή θα υπάρξει διαδικασία όχλησης κατά της πορτογαλικής ε, κυβέρνησης ε, λόγω ε, της, των διακρίσεων στην ισότητα και, της, και την ίση μεταχείριση αναλόγως με τη σύμβαση εργασίας κάθε κράτος, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Πορτογαλία στέλνουμε ένα μήνυμα σε άλλες χώρες και η Γαλλία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση κάθε πέντε χρόνια δηλαδή παραγράφονται όλα, ξαναρχίζουμε από το ε, σας το λέω βέβαια, εσείς θα έχετε ήδη πάει στη σύνταξη ενδεχομένως και μπορεί να μην σα αφορά το θέμα τότε, αλλά πραγματικά πρέπει να υπάρξει διαδικασία όχληση κατά τη Πορτογαλία προκειμένου να συμμορφωθεί οπωσδήποτε με το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ξέρω ότι προέρχεστε από ε, συνδικαλιστικό χώρο, κατάλαβα πάρα πάρα πολύ καλά την άποψή σας. Περνάμε τώρα στο επόμενο, στον επόμενο μιλητή, Πέτρου, θέλει να δώσεις τη θέση σου στην ε, κυρία Πιτέρα. Έχετε το λόγο, κυρία Πιτέρα. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Εγώ μια σύντομη ερώτηση έχω να κάνω προς τον εκπρόσωπο της Πορτογαλίας. Ε, ε το μελέτησα το πρόβλημα αυτό εντελεχώς και φαίνεται ότι έγινε μια μεταρρύθμιση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για το, το επιχείρημα στο νέο έγγραφο που παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι ο λόγος αυτού του εγγράφου, κύριε μαγιά. Κυρία Πρόεδρε, η περίπτωση αυτή που συζητούμε για την Πορτογαλία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Γίνεται μια κατάχρηση από πλευράς των κρατών σε σχέση με τη διαδικασία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Και ενώ ιδίω στα θέματα τη εκπαίδευση και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλύπτουν πάγιες και διερκείς ανάγκε, εν τούτη στα κράτη και στην περίπτωση αυτή η Πορτογαλία, αλλά σα λέω το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα, προτιμούν να έχουν συμβάσει ορισμένου χρόνου και κάθε έτος να τις ανανεώνουν τις συμβάσεις και αυτό γίνεται πρώτα απ' όλα διότι έτσι αμείβονται με μικρότερα ποσά οι εκπαιδευτικοί και δεύτερον γιατί τα κράτη δεν μπορούν να κάνουν ένα προγραμματισμό επειδή στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα και δικαίως βεβαίως στοιχίζουν οι εκπαιδευτικοί, επειδή τα κράτη, ιδίω η Ελλάδα, η Πορτογαλία και άλλα κράτη βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία μνημονιακή με περιορισμό των δημοσίων δαπανών και έτσι προτιμούν αυτές τις συμβάσεις γιατί λύνουν τα προβλήματά τους πρόσκαιρα. Μάλιστα σε ορισμένες χώρες αξιοποιούν και προγράμματα του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση αυτή. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία, δηλαδή εφόσον έχουμε συμβάσει ορισμένου χρόνου, ίδια πρόσωπα, πάγιε ανάγκε στου ίδιου χώρου, αυτέ οι συμβάσει μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Και είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία αυτή. Τέτοια προβλήματα είχαμε στην Ελλάδα, είχαμε πάρα πολλέ υποθέσει, είχαμε πάρα πολλά δικαστήρια και νομίζω ότι κάποτε πρέπει να λήξει αυτό. Και αυτό για να λήξει χρειάζεται οπωσδήποτε μία απόφαση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που να αναγκάζει την Πορτογαλία να συμμορφωθεί εν προκειμένου με τα ζητήματα αυτά. Και αντίστοιχε δραστηριότητε, αν υπάρχουν σε άλλα κράτη, πρέπει να ελεγχθούν. Τέλο, για να το ακούσει η Κομισιόν, είχα κάνει και μία ερώτηση που αφορούσε την Ελλάδα, όπου οι εκπαιδευτικοί που έχουν εργαστεί είχαν μια προπηρεσία. Και αυτή η προπηρεσία λαμβανόταν υπόψη για να ξαναπροσληφθούν την επόμενη χρονιά. Η Ελλάδα εντελώς παράνομα με μία εγκύκλιο φέτος δέχεται να αναγνωρίζει την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών από το διάστημα 2012-2014 αλλά δεν αναγνωρίζει την προϋπηρεσία τους το διάστημα 2010-2012. Αυτό είναι διακριτική μεταχείριση κατά πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με χρήματα του ΕΣΠΑ έχουμε παραβίαση και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό για να το ακούσει η Κομισιόν και να είστε βέβαιοι ότι σίγουρα και σύντομα θα έχετε μια τέτοια υπόθεση ενώπιον σας και από την Ελλάδα, διότι εδώ έχουμε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Excellent. Εξαιρετικά. Και τώρα θα δώσω το λόγο και πάλι στον αναφέροντα Ακούσατε τι είπαν οι συνάδελφοι από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Δύο λεπτά σας δίνω το λόγο. Thank you. Um, okay. uh, I see... Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Eu creio que daqui, se é que uh, me deu a entender, eu penso que... Από αυτό που κατάλαβα, νομίζω ότι ήδη έχουμε ένα θετικό μήνυμα. Αν κατάλαβα καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ξανανοίξει τη διαδικασία. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια νέα στοιχεία με συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς έχει κατάσταση από το 2014 μέχρι σήμερα, διότι συνέβη αυτό που σας είπα στο τέλος της παρουσίασή μας. Εξακολουθούμε να αποτελούμε αντικείμενο διάκρισης, και ακόμα και οι συνάδελφοι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, ε, συνάδελφοι που εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία και ε, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν μια κάποια αυτονομία. Μπορούν να προσλαμβάνουν ένα καθηγητή για πέντε χρόνια με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μετά μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να πάρει μέρος σε κάποιο διαγωνισμό και να πρέπει να αντιμετωπίσει συναδέλφους με 10-15 χρόνια εμπειρία. Επειδή όμω ο προηγούμενος έχει πέντε διαδοχικές αιτήσει ε, συμβάσεις, είναι αυτός που θεωρείται ότι προηγείται ε, στη διαδικασία του διαγωνισμού. Αν αυτό δεν είναι διάκριση, δεν ξέρω τι να σα πω, κρίνετε και μόνοι σας. Τώρα, ε, δεν κάνω σύγκριση με τους ε, ε, ανθρώπους που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου. Υπάρχουν ε, ε, συμβασιούχοι που εργάζονται για πέντε συναπτά έτη και όταν ε, υποβάλλονται, περνάνε από διαδικασία διαγωνισμού θεωρούνται ανώτεροι βαθμολογικά από τους άλλους και οι συνάδελφοι που εργάζονται 10-15 χρόνια και δεν έχουν ίσως ε, διαδοχικές συμβάσεις θεωρούνται με λιγότερη εμπειρία. Το κράτος όμως είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα όπως και εμείς ε, είναι ε, εργαζόμενοι που εργάζονται σε σχολικά ιδρύματα που υποστηρίζονται και αυτά από το κράτος. Δεν είναι αποκλειστικά ιδιωτικά. Υπάρχει χρηματοδότηση από το Πορτογαλικό κράτος και στήριξη από το Πορτογαλικό κράτος. Υπάρχουν συμβασιούχοι καθηγητές οι οποίοι μπορούν από εκεί και πέρα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με τις ίδιες προϋποθέσεις εμείς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσετε και πάλι το λόγο. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Εκφράσατε τις απόψεις σας. Και μου φαίνεται ότι θέλετε να μείνει η αναφορά ανοιχτή. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει τις πληροφορίες που θα μας δώσει μετά την αξιολόγηση των καινούριων στοιχείων. Έτσι καταλαβαίνω τα σχόλια των συναντέλφων στην παρούσα φάση. Συμφωνείτε? Ναι, πολύ ωραία. This is what we do then. Αυτά θα κάνουμε λοιπόν. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το 9, στην ημερήσια διάταξη. Μία σειρά αναφορών για την ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και κατά παραβίαση της συγκεκριμένη οδηγίας. Έχετε τα αριθμητικά στοιχεία μπροστά σας. Θα δώσω το λόγο στους ετούντες που εκπροσωπούνται εδώ από δικηγόρους. Θα μπορούσατε παρακαλώ να περιοριστείτε σε 2-3 λεπτά, γιατί μετά το 12.30 δεν θα έχουμε και τερμηνία. Και άρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν το διάλειμμα για μεσημεριανό. Σας παρακαλώ, σύντομη. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή και για τους συναδέλφους ασφαλώς. Έχετε το λόγο, Μάριο Ντινόσο. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής, ε, και πάλι θα συζητήσουμε επισφαλή σε θέση εργασία. Η Ιταλία τον Αύγουστο ενέκρινε νομοθεσία που θεωρείται ε, η νομοθεσία για τα καλά σχολεία, η οποία νομοθεσία συμπεριέλαβε τις υποδείξεις και θα μπορούσα να πω και τις συστάσεις ε, που επέβαλαν να γίνει προσαρμογή της Ιταλικής νομοθεσίας στις αρχές ε, του Ιταλικού Συντάγματος και ε, στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινοτικό δίκαιο, επιλύοντας εν μέρη το πρόβλημα των διδασκόντων. Εγώ παρεμβαίνω υπέρ της διαδικασίας στα δημόσια σχολεία για τη μονιμοποίηση του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε κάτι. Η νομοθεσία για το νέο σχολείο δεν κάνει καμία παρέμβαση για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Εξακολουθούν να έχουν επιφαλή θέσει εργασίας όπως συνέβαινε και πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Και ε, υπάρχουν, ε, όπως και ο κύριος Δηλούσο, πάρα πολλά ε, άτομα τα οποία εργάζονται για πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Δηλούσο εργάζεται για 11 χρόνια και υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που εργάζονται για 15-20 χρόνια ε, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εξαμηνιές, ετήσιες και ούτω καθεξής. Αυτό συνιστά κατάχρηση της ανανέωσης των συμβάσεων, διότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσει που ακούσαμε και από την προηγούμενη έκθεση ε, για την ε, πορτογαλική κατάσταση δεν ε, βασίζονται στις αντικειμενικές απαιτήσεις και τις αντικειμενικές ανάγκες και επομένως πρόκειται για κατάχρηση μιας κατάστασης η οποία εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα οδυνηρή και να δημιουργεί φυσικά προβλήματα στη ζωή αυτών των εργαζομένων που αποτελούν και αντικείμενο διάκρισης ενώπιον των μονίμων υπαλλήλων, αλλά και αντικείμενο διάκριση ε, ενώπιον των συναδέλφων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την Επιτροπή σας, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις που παρουσίασε η Ιταλική κυβέρνηση, που σε καμία περίπτωση δεν παρενέβη για να επιλύσει το πρόβλημα, δεν έχουν βοηθήσει και δεν έχουν ε, ε ρυθμίσει την κατάσταση αυτών των εργαζομένων, θα ήθελα να ζητήσω να ξανανοίξει η διαδικασία επιπαραβάση και να παρακολουθήσει την κατάσταση στην Ιταλία μέχρι να υπάρξει μια λύση ε, στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος στον αναφέροντα MR της 1302 αναφοράς. Δύο λεπτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι και εγώ αναφέρουσα και το 2010 ήμουν εδώ στην Επιτροπή σας. Να επαναλάβω κι εγώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα έκτοτε, διότι ο νόμος ε, για τα καλά σχολεία ε, ρυθμίζει μόνο το θέμα των διδασκόντων. Επομένως εμείς όχι μόνο αποτελούμε αντικείμενο διάκριση σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό, τώρα υπάρχει και διάκριση σε σχέση με τους ε, συμβασιούχους διδάσκοντες. Πρόκειται για περαιτέρω διάκριση που τιμωρεί ακόμα και περισσότερο το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξής. Εμείς και προσωπικά, προσωπικά ε, προσφύγαμε στα δικαστήρια ώστε να αναγνωριστούν τα δικαιώματά μας και να προστατευτούμε κάπως, αλλά δυστυχώ, ε, στην Ιταλία ή τουλάχιστον στην περιοχή της Κατάνια από την οποία κατάγομαι εγώ, τα δικαστήρια πάντα αναβάλουν τι υποθέσει μας. Ε, στην αρχή περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου, κάποια στιγμή είχαμε επιτέλους αυτή την απόφαση και τώρα τα δικαστήρια αναβάλουν ε, συνεχώς το θέμα και δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα γιατί περιμένουμε την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Εδώ και πέντε χρόνια λοιπόν περιμένουμε, δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα πρέπει να περιμένουμε, προκειμένου να μας παρασχεθεί έστω μια ελάχιστη προστασία. Εσείς λοιπόν ως πολιτικοί ε, θα πρέπει να κάνετε κάτι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μία προστασία ε, από δικαστικής πλευράς. Και μας μας ε, στεναχώρησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι έκλεισε η διαδικασία επί παραβάση, γιατί υπήρχε διαδικασία επί παραβάση και για το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Το μόνο που άλλαξε είναι για το διδακτικό προσωπικό και όχι για μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήσασταν και τόσο σύντομοι. Και τώρα ο λόγος ε, στην κυρία Λορέντσα Λοκάστη. Καλημέρα σας είμαι εκπρόσωπος της κυρίας Βαλέρια Πιτσάρη, που είναι και αυτή συναδελφός μου, και είμαι και εγώ ε, συμβασιούχος ε, με επισφαλή θέση εργασίας εδώ και 15 χρόνια. Πρέπει να πω το εξής. Εγώ, όπως και η συνάδελφος, όχι μόνο λαμβάνω συμβάσεις από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 1η Αυγούστου και το αντίθετο, εγώ είχα συμβάσεις για 7 διαδοχικά χρόνια και έκανα και διάφορες αναπληρώσεις, οι οποίες και αυτές ήταν διαδοχικές. Αυτό όμως το οποίο με εκπλήσει είναι ότι κάθε χρόνο η Ιταλική κυβέρνηση επινοεί νέα περίεργα πράγματα. Για παράδειγμα, την κινητικότητα των εργαζομένων των σχολείων, γιατί ε, χρησιμοποιούν ε, ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και λαμβάνουν ε, θέσεις ε, δικές μας, διοικητικού προσωπικού. Επίσης, ακατάλληλους διδάσκοντες. Υπάρχουν διδάσκοντες που δεν είναι κατάλληλοι να διδάσκουν σε τάξη και τους βάζουμε σε κάποια διοικητική θέση που σημαίνει ότι αφαιρείται μια θέση σε εμά του συμβασιούχου. Το τελευταίο δε επινόημα της κυβέρνησης είναι ε, τους, ε, ε, το πλεονάζον προσωπικό των ε, περιφερειών. Πού θα τους πάμε, θα τους πάμε να δουλέψουν το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, γιατί αυτοί όχι μόνο έκαναν αυτό το νέο σχολείο και τη νέα νομοθεσία και έχουν προσλάβει νέους διδάσκοντες, αλλά έχουν μπλοκάρει και εμάς. Γιατί για μας... Τώρα αυτό που κάνουν είναι αναγνώριση του προσωπικού του σχολείου και δεν έχουν αποδεχτεί πουθενά ότι υπάρχουμε κι εμείς. Μάλιστα στην Ιταλία έχουν ε, αναστείλει τους αναπληρωτές, ε, δεν χρησιμοποιούν τους διοικητικούς ε, βοηθούς και έχουν περιορίσει πάρα πολύ τα δικά μας τα καθήκοντα. Εγώ εργάζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γερνάω μαζί τους, γερνάω με όλες αυτές τις αλλαγές και πραγματικά με κουράζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, δεν είναι ζωή αυτή και δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα. Grazie, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι εδώ εκ μέρους του κυρίου Τζουζέπε Ρουμόρε Παγκάνο. Όταν υπέβαλε και τις δύο αναφορές το 2013 και το 2012, ο ε, κύριος Παγκάνο ήταν ε, συμβασιούχος, αλλά ε, στο μεταξύ προσελήφθη χάρη σε κάποιες κενές θέσεις ε, στη διάρκεια του ε, σχολικού έτους και χάρη στο turnover. Και δυστυχώς όμως, όπως εξήγησαν αρκετοί από τους προηγούμενους, πρόκειται για μια εξαίρεση, γιατί η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε μεν να δώσει μια λύση στις διαδικασίες επιπαραβάσεων παραβάση που ξεκίνησε η Επιτροπή σας, αλλά καθορίζοντας μόνο εξαιρετικό πλάνο προσλήψεων, μόνο για τους διδάσκοντες, ενώ για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δεν έχει προβλέψει τίποτα. Δεν έχει προβλέψει ούτε ένα σχέδιο προσλήψεων, ούτε κάποιες προσλήψεις οι οποίες ε, θα ε, ε, είναι διαδοχικές. Προέβλεψε απλώς τελείως διαφορετική αλλαγή στο ρόλο τους, έχει αφήσει κάποιες κενές θέσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν κανονικά ε, στους ε, συμβασιούχους ε, αυτούς που εργάζονται σε, ως διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Τώρα έχει προβλέψει κινητικότητα για το πλεονάσμα προσωπικό των περιφερειών και τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζει μια μεταρρύθμιση που ασχολείται με την εξωτερική ανάθεση των διοικητικών ε, θέσεων στα σχολεία, επομένως θα αφαιρέσει περισσότερες θέσεις σε αυτούς τους συμβασιούχους. Επομένως η Ιταλική κυβέρνηση έχει προβλέψει να βοηθήσει μόνο τους διδάσκοντες και έχει κάνει προβλέψεις για την επόμενη χρονιά μόνο για τους διδάσκοντες. Γιατί δεν έχει προβλέψει κάτι αντίστοιχο για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ούτε για φέτος, ούτε για την επόμενη χρονιά. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή σας να ξανανοίξει τη διαδικασία επιπαραβήση, ζητώντα από την κυβέρνηση να προβλέψει ένα σχέδιο προσλήψεων Λοιπόν και για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί και αυτοί εδώ και 10 χρόνια έχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας και τους αξίζει να λάβουν αντίστοιχες προϋποθέσεις όπως και οι διδάσκοντες. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Merci, Madame la Présidente. Également Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά ανέλαβε τα ενία αυτή τη υπόθεση από τι εκατοντάδε καταγγελίε που λαμβάνει από το 2009 και εξή για το θέμα αυτό. Και πρέπει να πω ότι σήμερα ε, κατόπιν νέα συνδικαλιστική εκστρατεία ε, λαμβάνουμε πάνω από ε, χίλιες καταγγελίες, κάτι ε, το οποίο πραγματικά μας δημιουργεί πολλές προκλήσεις και σε μας και στη μεταφραστική υπηρεσία. Κατόπιν των καταγγελιών αυτών ε, εκτιμήσαμε ότι στο παρελθόν το σύστημα που αφορά το, τις συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν συμμορφώνονταν με την οδηγία και όπως κάναμε και για την Πορτογαλία ξεκινήσαμε διαδικασία όχλησης κατά των εθνικών αρχών της Ιταλίας. Επίσης, δρομολογήσαμε μία διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ιταλίας. Πρέπει να πω απλώς για να διευκρινιστεί γιατί νομίζω ότι θα ξανατεθεί το θέμα κάποια στιγμή στην Επιτροπή σας. Υπάρχουν καταγγελίες ε, στο ε, πλαίσιο των σχολείων αλλά υπάρχουν και, υπάρχουν και εκατοντάδες καταγγελίες ε, για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα της Ιταλίας. Αν ολοκληρώσαμε την διαδικασία για το σχολικό ε, πλαίσιο υπάρχουν καταγγελίες που θα παραμείνουν ανοιχτές για το υπόλοιπο του δημοσίου τομέα στην Ιταλία. Αυτό θα ήθελα απλώ να το διευκρινίσω. Δεν θα υπενθυμίσω μόνο αυτό που λέει και που δεν λέει η οδηγία για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πάντως το πρίσμα της ανάλυσης μας παραμένει το ίδιο. Αν μία από τις ρήτρε ε, κατά των καταχρήσεων ε, ενεργοποιηθεί, είναι αυτό αρκετό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δεχθεί ότι το σύστημα, το εθνικό, είναι πλέον συμβατό. Και στο πλαίσιο αυτό ε, λάβαμε και όχι μόνο εμείς αλλά και οι καταγγέλλοντες και τα συνδικαλιστικά κινήματα ε, και ε, οι βουλευτές στην Ιταλία για, την, για, το, για τα Ιταλικά σχολεία ε, ότι θα ε, γίνουν προσλήψεις ε, μόνιμου προσωπικού πλέον για τους ανθρώπους αυτού και οι διαδοχικές συμβάσεις περιορίζονται στους 36 μήνες, ακόμη και αν δεν είναι διαδοχικές οι συμβάσεις και αποζημίωση για περιπτώσεις διαφορετικής μεταχείρισης μεταξύ συμβασιούχων μονίμου, περιορισμένου και ορίστου χρόνου θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ενωσιακή νομολογία είναι πάρα πολύ γνωστή σε σχέση με το θέμα της μονιμοποίησης και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών και των αναφερόντων ε, στην ε, παράγραφο 65 της υπόθεσης Φαμέγκο που αφορά συγκεκριμένα την Ιταλία και υπενθυμίζει στις εθνικές δικαιοδοσίες και στα εθνικά κοινοβούλια ότι έχει πολλές φορές τονίσει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ε, μονιμοποίησης για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που να προέρχεται, να προκύπτει από την οδηγία αν ένα από τα τρία μέτρα που περιέγραψα ε, προηγουμένως ε, αναλυφθούν. Τώρα, ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες εκστρατείες ε, ε, μονιμοποίησης που αφορούν ειδικότερα τους καθηγητές, όμως επειδή υπάρχει περιορισμός των 36 μηνών όπως σας είπα, αυτός, αφορά, αυτός ο περιορισμός αφορά όλο το προσωπικό του ε, σχολείου. Μιλάμε για το άρθρο 131 ε, της Ιταλικής νομοθεσίας, όπου αναφέρεται ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2016 οι συμβάσει ορισμένου χρόνου που έχουν συναυθεί με προσωπικό, διδακτικό, εκπαιδευτικό, κατάρτισης ε, και άλλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτήν τη μέγιστη περίοδο των 36 μηνών συμπεριλαμβανομένων ε, των ε, μη διαδοχικών συμβάσεων. Ε, η αποζημίωση σε περίπτωση διαφορετικής μεταχείρισης που προβλέπει η Ιταλική νομοθεσία ε, επίσης υπάρχει πλέον για το, για το διδακτικό προσωπικό. Γι' αυτό ακριβώς στο πλαίσιο της ανάλυσης του σχολικού τομέα ε, αποφασίσαμε αυτά που σας εξήγησα συγκεκριμένα με την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα κυρία Τζέα. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι αναπληρωτής εδώ στην Επιτροπή, αλλά είμαι πλήρες μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η οδηγία 1999 κάθετος 70, η οποία πλέον είναι 15 ετών, προέβλεπε δύο υποχρεώσεις, οι οποίες έπρεπε να ε, τηρηθούν απολύτως. Το γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος θα έπρεπε να καταδικάζει τις περιπτώσεις κατάχρησης και κάθε κράτος ε, θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από συγκεκριμένες κυρώσεις βάσει των οποίων θα τιμωρεί τις περιπτώσεις της κατάχρησης. Αυτές ήταν οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις που αυτή τη στιγμή δεν έχει εφαρμόσει η Ιταλία και γι' αυτό και ξεκίνησε μια διαδικασία επιπαραβάση. Γι' αυτό και υποχρεώθηκε η Ιταλία να νομοθετήσει και να κάνει το νόμο για αυτό το καλό σχολείο. Ε, υπάρχουν δύο λοιπόν ε, αυστηρά μέτρα. Η κυβέρνηση Ρέντσι ε, έκανε αυτή τη νέα μεταρρύθμιση για το καλό σχολείο. Αλλά έχει παραμείνει το πρόβλημα, διότι το άρθρο το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 131 παράγραφος ε, της νομοθεσίας για το καλό σχολείο, που λέγεται ότι οι συμβάσεις ε, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη διάρκεια των 36 μηνών, δεν καθορίζει ποιε είναι οι σχετικέ κυρώσει. Επομένω, επ' αυτή τη βάση, εμεί θα προτείνουμε και πάλι να γίνει μια επαλήθευση και να ανοίξει η διαδικασία επί παραβάση, διότι οι υποχρεώσει που έπρεπε να αναλάβει η νέα μεταρρύθμιση δεν έχουν τηρηθεί. Thank you very much. Κύριε Πρόεδρε, ε, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα από ό,τι φαίνεται και στην Ιταλία, διότι η τακτική είναι ίδια. Η αξιοποίηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου προκειμένου να μην υπάρχει μόνιμη απασχόληση. Μάλιστα, όπως είπαν και οι αναφέροντες, πάμε και σε μια διαδικασία πλέον αναδιάρθρωσης. Αυτή η κινητικότητα η οποία υπάρχει και θίγει τους ίδιους εργαζόμενους και θα έλεγα ότι και στην Ελλάδα είχαμε τα στοιχεία αυτής της κινητικότητας ήταν ένας τρόπος με τον οποίο οι δανειστές ήθελαν να περιορίσουν το προσωπικό στο δημόσιο και στην εκπαίδευση. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στις εργασιακές σχέσεις, ιδίως στο θέμα της εκπαίδευσης. Υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει στην Πορτογαλία, το είδαμε πριν, υπάρχει στην Ιταλία. Και πιθανόν να έχουμε και άλλες καταγγελίες. Θα έλεγα λοιπόν μήπως θα πρέπει η Επιτροπή μας να δει σφαιρικά αυτό το ζήτημα, Δηλαδή να εξετάσουμε όλες μαζί αυτές τις περιπτώσεις που αφορούν ε, κράτη ε, τα οποία δεν εφαρμόζουν σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ε, αξιοποιούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενώ στην πράξη πρέπει να έχουμε συμβάσεις αορίστου χρόνου και μήπως πρέπει να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, μήπως πρέπει να ετοιμάσουμε ίσως και μια ερώτηση στην ίδια την Επιτροπή για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα της απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην εκπαίδευση σε πολλά κράτη. Ας δούμε λοιπόν στοιχεία και από άλλες αναφορές, να μας βοηθήσει εδώ και η γραμματεία. Μπορεί να έχουμε και άλλες αναφορές οι οποίες είναι σε εξέλιξη και αναμένουν, ούτως ώστε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το ζήτημα αυτό. Ως πρόταση για παρέμβαση της ίδιας της Επιτροπής. Και για το θέμα της Ιταλίας νομίζω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτό για να δούμε πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί πραγματικά η νομοθεσία ε, σε σχέση με τις περιπτώσεις που μας ανέφεραν οι συνάδελφοι και που από ό,τι φαίνεται κινδυνεύουν και με απόλυση διότι πιθανώς στη θέση τους το τεχνικό προσωπικό να μπουν κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες από ό,τι φαίνεται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές χώρες και όχι μόνο στην Ιταλία ή στην Πορτογαλία ή στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Δίνω το λόγο στον κύριο Μαρτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ πιο σύντομα θα μιλήσω από ό,τι πριν, ελπίζω. Πάντως θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος Μαριάς. Ε, το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι εγκάρσιο. Πρέπει εκείνη να μας εξηγήσει τι είναι η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μπορεί να αφορά, ε, για παράδειγμα, την αντικατάσταση ενός υπαλλήλου που ασθενεί τούτων λεχθέντων όμως ε, Χαίρομαι πολύ που υπάρχει εδώ μία εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι Μεσένος θα αντιταχθεί στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Όμως, από ποια, λογική, από ποια στιγμή και μετά υπάρχει όχληση κατά μίας ε, χώρας ε, ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο επιβάλλεται για να μπορέσει να συμμορφωθεί το κράτος μέλος. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν 15, 10 χρόνια, 5 χρόνια, αναφέρονται σε εδώ και πολύ καιρό. Περιμένει ο κόσμος. Πόσο θα περιμένουμε. Η Πορτογαλία και η Ιταλία μπορούν να καθυστερούν και άλλα χρόνια. Και μια τελευταία παρατήρηση γιατί ξέρω ότι γίνεται και εδώ και θα επανέλθουμε με μια αναφορά για το προσωπικό μας εδώ. Εάν ποτέ ε, σας δίνει, αν ποτέ αν ποτέ σας δώσουν μια επιλογή αλλαγής του, ε, του, της σύμβασής σας, εύχομαι να μην πέσετε σε μια, κακή συνέ, ε, σε μια κακή κυβέρνηση που θα σας δημιουργήσει τα χειρότερα προβλήματα. Πρόεδρος, ε, βλέπω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων εδώ, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω αν είναι απολύτως απαραίτητο να πάρετε το λόγο, να πάρετε το λόγο, αλλά αλλιώ παρακαλώ να απόσχετε. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα απλώ να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπαν σαφέστατα οι συνάδελφοι, ότι πρόκειται για ένα συστημικό πρόβλημα. Νομίζω ότι ε, φάνηκε αυτό και από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κράτη-μέλη, σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε στην Ιταλία και η Ιταλία ε, επανειλημμένος ε, κάνει κάποιες ε, διαδικασίες συγκάλυψης για να αποφύγει τη διαδικασία επί παραβάση και προσπαθεί να βάλει ένα βούλωμα, σε ένα ε, τσιρότο σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ανακύπτει συνεχώς, είναι κάθε χρόνο φρικτά τα προβλήματα και η Ιταλία κάθε χρόνο δεν κάνει τίποτα για να επιλύσει συγκεκριμένα το πρόβλημα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονό ότι αυτό γίνεται συστηματικά. Είναι διαδικασίε επί παραβάση και πολύ συχνά με μία απλή απόφαση ή ένα διάταγμα, μια μικρή μεταρρύθμιση, προσπαθούν να σταματήσουν τη διαδικασία επί παραβάση. Και μετά από του ελέγχου που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι η παράβαση συνεχίζεται. Το βλέπουμε και με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Η Ιταλία. Ε, έχει συνέχεια περιφερειακά σχέδια για την επίλυση του προβλήματος και τελικά το πρόβλημα δεν λύνεται. Αυτό λοιπόν ε, είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εδώ στο Κοινοβούλιο. Thank Ευχαριστώ. Να στραφώ τώρα προς τις αναφέρουσες και να ρωτήσω αν θέλετε να κάνετε ένα τελικό σχόλιο. Έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο μία παρατήρηση στα όσα είπαμε και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή σας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η υποστήριξη της Επιτροπής. Το να επαφιόμαστε μόνο στο δικαστικό σύστημα δημιουργεί περαιτέρω διακρίσει. γιατί κάθε δικαστή στην Ιταλία είναι ανεξάρτητο και η ίδια υπόθεση αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Βέβαια αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί όλε οι διαδικασίε εν αναμονή τη απόφαση του δικαστηρίου, μετά είχαμε την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου, ακόμα δεν έχει διορίσει δικαστέ το συνταγματικό δικαστήριο για πολιτικού λόγου. Επομένω, θα ήθελα να το υποστηρίξετε αυτού του εργαζομένους, γιατί ίσω, εάν υπάρξει ασφάλεια δικαίου θα μπορέσει ε, το, να βελτιωθεί η κατάσταση και το κράτος να μην καταχράται την ίδια του την νομοθεσία. Ε, αυτό θα πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρόλα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, από το νόμο για το καλό σχολείο είχε προβλεφθεί ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν στους 36 Μήνε, αλλά δεν έχει προβλεφθεί καμία κύρωση. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει να υποστηρίζει αυτού του επισφαλείς εργαζομένους, ε, ε, θα μπορέσει να υπάρξει κάποια συνέχεια ε, και αλλιώ ελοχεύει ο κίνδυνο να χάσουν τι δουλειέ του αυτοί οι άνθρωποι και η Ιταλική κυβέρνηση θα κάνει διαγωνισμού μόνο για του διδάσκοντε και θα αποκλείσει τελείω το, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Επομένω, δεν θα μπορούν να έχουν μια σύμβαση εργασία, απλώ και μόνο γιατί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων και δεν είναι διδάσκοντε. Επομένω, θα ήθελα να σα ζητήσω να του βοηθήσετε ώστε η Ιταλία να αναγκαστεί να παρέμβει και για αυτό το προσωπικό. Σας ευχαριστώ πολύ και με αυτό ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών για σήμερα. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα πρέπει να μην ανοιχτεί αυτή η υπόθεση, νομίζω. Να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ε, συνεχίσει να εξετάζει την κατάσταση στην Ιταλία και να μας ε, ενημερώσει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το στοιχείο της διακριτικής μεταχείρισης όπως ε, διατείνονται οι αναφέροντες. Γιατί η διακριτική μεταχείριση είναι ενάντια στις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοι από ό,τι κατάλαβα θέλουν να μπει το θέμα αυτό στην συνεδρίαση των συντονιστών για να αποφασίσουμε κατά πόσον θα υπάρξει προφορικό ερώτημα για την οριζόντια προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε σχετική απόφαση τώρα. Θα πρέπει να την πάρουν την απόφαση οι συντονιστέ. Αυτό όμω προτείνω για τη συνέχεια για το θέμα αυτό. Κάτι άλλο, κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε ή θα μπορούσαμε να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Πολύ σα ευχαριστώ και τώρα Σα εύχομαι καλό διάλειμμα. Τα λέμε το απόγευμα. Ευχαριστούμε και του αναφέροντε που παρευρέθησαν.